προκειμένου να εξασφαλιστεί το δικαίωμά τους για δίκαιη δίκη και μάλιστα χωρίς ε, δικαιολόγητη χρονοτριβή. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε κυρία Επίτροπε Νταμανάκη και κλείνοντας ε, κατατεθήκαν έξι, ε, έξι ψηφίσματα. Η ψηφοφορία ακολουθεί σε λίγο. Περνάμε λοιπόν στις ψηφοφορίες. Ε, καταρχάς έξι ψηφίσματα σε ό,τι αφορά την κατάσταση στο Μπαγκλαντές. Η συνάδελφος Λόχ Μπίλερ, διαδικαστικό. Θα ήθελα να διορθώσω ένα ασφάλμα σε ό,τι αφορά τα περιστατικά. Θα ψηφίσουμε το ψήφισμα για τον ε, Μπαγκλαντές, αλλά στο AI αναφέρεται μετά τις εκλογές το 2001 και το 2005. Δεν έλαβαν χώρα εκλογές το 2005, γι' αυτό θα θέλαμε να διαγράψουμε το 2005 πρώτο ψηφίσουμε. Ευχαριστώ. Θα μπορούσατε να το σημειώσετε. Δεν ξέρω αν υπάρχουν ε, ε, αντιρρήσεις, ενστάσεις κατά της προφορικής τροπολογίας. Μάλιστα, ωραία. Ψηφίζουμε λοιπόν την παράγραφο 4 του αρχικού κειμένου. Ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Μετά την παράγραφο 13, τροπολογία 1, με ονομαστική κλίση, έναρξη ψηφοφορίας, παρακαλώ. Συνάδελφε, time. Για, συγγνώμη, Πήρα μία νέα κάρτα ψηφοφορίας πριν από λίγο, αλλά δεν λειτουργεί. Πατάω το θετικό πρόσημο, αλλά δεν μετριέται η ε, ψήφος μου. Δεν προλαβαίνω να παναφέρω άλλη κάρτα. Δεν λειτουργεί και στη διπλανά ε, έδρανα. Δεν ξέρω γιατί. Συνάδελφε, μήπως έχετε αφήσει την παλιά σας κάρτα κάπου αλλού και γι' αυτό δεν λειτουργεί η καινούργια όπως και να έχει ανοιχτή ακόμα η ψηφοφορία, πέρας ψηφοφορίας τώρα. Μπορούμε να κλείσουμε την ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Και σημειώνουμε και την ψήφο της κυρίας Τέιμ. Και περνάμε τώρα στην αιτιολογική σκέψη I, έτσι όπως τροποποιήθηκε. Συμφωνείτε, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Και τώρα περνάμε στην τελική ψηφοφορία για το τροποποιημένο ψήφισμα. Με ονομαστική κλίση, έναξη ψηφοφορία, παρακαλώ. Αν ψήφισατε όλοι, κλείνει η ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Και περνάμε τώρα στην ε, ψηφοφορία για ε, έξι ψηφίσματα σε ό,τι αφορά το Ιράκ και την δραματική κατάσταση των μελλοντικών ομάδων. Έχουμε ένα κοινό ψήφισμα πέντε ομάδων, την οποία θα ψηφίσουμε. Παράγραφος 6, υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Παράγραφος 7. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Μετά την παράγραφο 10 έχουμε τροπολογία 1. Υπέρ. Κατά. Να το ελέγξουμε παρακαλώ έναρξη ηλεκτρονικής ψηφοφορίας. Αν ψηφίσατε όλοι, πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα, μετά την παράγραφο 10, είναι η τροπολογία 2 των πρασίνων υπέρ. Κατά. Και αυτό θα ήθελα να το ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Έναρξη ψηφοφορίας, παρακαλώ. Αν ψηφίσετε όλοι, πέρας. Απορρίπτεται επίση στο Β σε δύο τμήματα παρακαλώ. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. απόχέ. Εγκρίνεται. Και τώρα περνάμε στην τελική ψηφοφορία για το τροποποιημένο κείμενο του ψηφίματος με ονομαστική κλίση. Έναξη ψηφοφορία, παρακαλώ. Να ψηφίσετε όλοι. Πέρας ψηφοφορίας με μία αποχή ομόφωνη έγκριση του ψηφίσματος. Τώρα, ψηφοφορία για πέντε ψηφίσματα για την περίπτωση του Αραφάτ Τζαραντάτ και την κατάσταση των Παλαιστινίων κρατουμένων στις Ισραηλινές φυλακές. Έχουμε καταρχάς το ψήφισμα του ΕΛΚ να ψηφίσουμε με ονομαστική κλίση το ψήφισμα αυτό. Έναρξη ψηφοφορίας παρακαλώ. Ψήφισατε όλοι. Πέρα ψηφοφορία. Απορρίπτεται με ισοψηφία. Και τώρα περνάμε στο κοινό ψήφισμα τεσσάρων ομάδων. Καταρχά, παράγραφο 5 του αρχικού κειμένου σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα, παρακαλώ, υπέρ. Κατά. Αποχές. Έγκρινεται. Δεύτερο τμήμα, υπέρ κατά για να ψηφίσουμε παρακαλώ ηλεκτρονικά το δεύτερο τμήμα της παραγράφου 5 για να ελέγξουμε. Είναι οριακή. Οριακό το αποτέλεσμα. Ψήφισατε όλοι. Πέρας ψηφοφορίας παρακαλώ. Εγκρίνεται. Παράγραφος 8 του αρχικού κειμένου σε τρία τμήματα. Πρώτο τμήμα παρακαλώ υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. και εδώ παρακαλώ να το ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Έναρξη ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρασε. Έγκρινεται. Τρίτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές η ίδια ψηφοφορία, η ίδια πλειοψηφία. Αν θέλετε το ελέγχουμε. Ελέγχουμε το τρίτο τμήμα της παραγράφου 8, παρακαλώ ηλεκτρονικά. Έναρξη ψηφοφορίας. Ψηφίσατε όλοι. Πέρασε. Μεγαλύτερη πλειοψηφία ακόμα. Παράγραφος 10, σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Ας το ελέγξουμε και αυτό ηλεκτρονικά έναρξη ψηφοφορίας. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Παράγραφος 11 του αρχικού κειμένου υπέρ. Κατά. Να το ελέγξουμε και αυτό παρακαλώ να, ψη... ελέγξουμε ηλεκτρονικά την παράγραφο 11. Ψήφισατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται επίση. Και τώρα περνάμε στην τελική ψηφοφορία για το τροποποιημένο κείμενο. Έναρξη ψηφοφορία, παρακαλώ. Haben Ψηφίσατε όλοι. Πέρα ψηφοφορία. 32 ψήφοι υπέρ, 29 κατά, εγκρίνεται. Και έτσι ολοκληρώσαμε την συνεδρίαση. Τα πρακτικά θα τα λάβετε για έγκριση στην επόμενη, για την επόμενη σύνοδο. Και τα ψηφίματα τα οποία εγκρίθηκαν θα α, διαβιβαστούν στους υπεύθυνους.